Kollegen? Ε? ja. so, dear colleagues, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω, παρακαλώ, βάλτε και τα ακουστικά σας, γιατί μια και έχουμε τις υπηρεσίες τις γλωσσικές στη διάθεσή μας, σκοπεύω να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους Κάποια ακόμη περιμένουμε να φτάσουν. Να κάτω φτάσουν. Έχουμε και κάποιους ολίγους εκπροσώπους του ΕΛΚ, ολίγους δυστυχώς, διότι είχε στο Παλέρμο μια συνεδρίαση το ΕΛΚ, από ό,τι γνωρίζω. Δυστυχώς λείπουν πολλοί συνάδελφοι. Από ό,τι όμως έμαθα, ο κύριος Πίτη Κάικ, ναι, να ναι, έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει και εκείνος. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε ως εκ τούτου, πιστεύουμε, μια ικανοποιητική εκπροσώπηση του ΕΛΚΑ. Α, και τενούτα είναι εδώ. Καλώ ήρθε. Όσο πιο πολλού εκπροσώπου έχουμε, τόσο καλύτερο. Και θα ήθελα να συστήσω τώρα τις ε, τροπολογίε που έχουν προτεθεί στην ε, έκθεση. Παρακαλώ λοιπόν πρώτα την Περβάν Μπερές, μια κοινή συντάκτρια αυτής της ε, έκθεση των συμπερασμάτων να ε, κάνει την παρουσίαση των τροπολογιών και τα σχόλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις 522 τροπολογίες που είχατε την καλοσύνη να καταθέσετε για την έκθεση αυτή. Η αντίδρασή μου για τις τροπολογίε αυτές ήταν διπλή και θετική και αρνητική. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή βάση για συμβασμό. Ήταν θετική η αντίδρασή μου από την άποψη ότι είδα μια πολύ πιο ομοιόμορφη, μια πολύ πιο ομοιογενή προσέγγιση που σέβεται το πνεύμα της συμφωνίας μας που κατέληξε στο ψήφισμα της 20ης ε, Οκτωβρίου του 2010 και με τα χρονικά περιθώρια που είχαμε και μας υποχρεώνουν να υιοθετήσουμε την τελική έκθεση στην Ολομέλεια ταυτόχρονα, στην ίδια Ολομέλεια δηλαδή με την ε, έγκριση της έκθεσης και της Επιτροπής ΣΟΥΡ θα γίνουν σεβαστά κατά πάσα πιθανότητα αυτά τα χρονικά περιθώρια μετά από τις ε, τροπολογίες που καταθέσατε. Παρ' όλα αυτά, εγώ ελπίζω ότι θα ήταν λιγότερες τρυπολογίες και δεν θα κατακλυζόμουν αυτή την πληθώρα. Πολλό δε μάλλον που μεταξύ μας είχαμε συμφωνήσει και σε ένα κανόνα. Είχαμε συνεννοηθεί οι τροπολογίες να υποβάλλονται μόνο υπό την αιγίδα των συντονιστών ή των σκιωδών εισηγητών. Συγκεντρώνοντα φυσικά και άλλε υπογραφές. Από τις 500 όμως 22 τροπολογίες που συνολικά κατατέθηκαν, μόνο 313, δηλαδή το 66% του συνόλου ε, τηρούν αυτόν τον κανόνα. Λυπούμε ειλικρινά, γιατί εγώ ήμουν υπέρ αυτού του κανόνα που είχαμε κανονίσει και θεσπίσει μεταξύ μας. Έτσι υπάρχει μία ανισότητα από την αρχή, όπως ε, και κατά την έναρξη αυτής της περίοδου κρίσης. Και διαπιστώνω ότι μερικοί συνάδελφοι είναι πολύ πιο πειθαρχημένοι σε ό,τι αφορά την τήρηση αυτού του κανόνα. Οι πράσινοι είχαν το πρώτο βραβείο, γιατί δεν υπέβαλαν καμία επιπλέον τροπολογία από τις αρχικές ε, υπό την αιγύδα του συντονιστή τους. Μετά τη δεύτερη θέση κέρδισε η δική μου πολιτική ομάδα, που με μόνο δύο τροπολογίες ε, εκτός συνολικής ε, συμφωνίας κατέθεσε. Δεν πρόκειται τώρα να ταξινομήσω με βάση αυτές τις επιδόσεις όλες τις πολιτικές ομάδες. Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι οι φιλελεύθεροι θα μπορούσαν να είχαν και καλύτερες επιδόσεις, γιατί από τις 89 τροπολογίες μόνο οι 59 τροπολογίες τους εμπίπτουν στον κανόνα της ε, συνυπογραφής με το συντονιστή. Ενώ στο ΕΛΚ από των 60 τροπολογίες, 60 μόνο έχουν υπογραφεί από το συντονιστή τους. Οι 60 τροπολογίες που έχουν ε, συνυπογραφεί από το συντονιστή του ΕΛΚ μου δίνουν κάποιες ελπίδες ε, για ενδεχόμενο συμβασμό, συμβαστική λύση με το ΕΛΚ. Μεταξύ μας πάντως και για όσους ε, συμμετείχαν στις εργασίες της Επιτροπής με αφοσίωση, ο κανόνας ήταν σαφής εξ αρχής. Οπότε, ε, κατά τη ε, διαμόρφωση συμβεστικής λύσης, ε, αισθάνομαι την, το καθήκον να ευνοήσω αυτούς που τήρησαν τον κανόνα και αυτούς που υπέβαλαν υπό την αιγύδα του συντονιστή τους και με συμφωνία του συντονιστή τους στις τροπολογίες και για τις υπόλοιπες θα ενεργήσω κατά το δοκούν. Αλλά δεν αισθάνομαι δεσμευμένη, υποχρεωμένη να λάβω υπόψη όλες αυτές τις επιπλέον τροπολογίες. Είναι ασθενιστό τις απόψεις που παρουσιάζουν. Μάλιστα για 32 τροπολογίες του ΕΛΚ από ό,τι κατάλαβα και θα τις αναφέρω και ονομαστικά τις τροπολογίες ε, των κυρίων Σαρή και Σάγια και 15 τροπολογίες, για 15 τροπολογίες των φιλελευθέρων, δημοκρατών και φιλελευθέρων του κυρίου Καρλ Χάγκλουντ Πρόκειται για καταστάσεις που αφορούν την εσωτερική τους, ε, για που αφορούν την ε, εσωτερική της πολιτική κατάσταση και νομίζω ότι δεν έχουν πια αντικείμενο αυτές οι τροπολογίες γιατί η κατάσταση έχει ξεπεραστεί. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ καλή χειρονομία εκ μέρου του να αποσύρουν αυτέ τι τροπολογίε που είναι πια παροχημένε. Για του φιλελεύθερου ήθελα να πω ότι οι τροπολογίε του κ. Καρλ Χάγκλουντ που από ό,τι βλέπω απουσιάζει σήμερα το απόγευμα. Οι τροπολογίες αυτές ε, επαναλαμβάνουν πιστά τις ε, τροπολογίες που έχει καταθέσει ο συντονιστής των φιλελευθέρων εκ μέρους ε, του συνόλου της ομάδας. Αυτά ως προς το τυπολατρικό γραφειοκρατικό τμήμα και το πιο βαρετό της συζήτησης. Τώρα ως προς την ουσία. Τρεις γενικές προκαταρκτικές παρατηρήσεις πριν επισέλθουμε σε πιο διεξοδική ανάλυση. Πρώτη γενική παρατήρηση αφορά τις τροπολογίες που ζητούν την ε, πανεισαγωγή της φορολογίας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε διάφορα σημεία της τελικής έκθεσης της έκθεσης κρίσης της Επιτροπής μας. Γνωρίζετε τη θέση μου για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και μάλιστα την ψηφίσαμε στην πρώτη έκθεση της Επιτροπής Κρίς και μάλιστα η θέση αυτή επιβεβαιώθηκε και με την στάση που πήραμε εγκρίνοντα την έκθεση κυρία Ποδηματά. Κατά τη γνώμη μου ήταν αυτή η καλή βάση και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεταξύ μας συμφωνούμε ε, για ορισμένα σημεία, αν μεταξύ μας συμφωνήσουμε για την επανεισαγωγή αυτού του φόρου επί το χρηματοπιστωτικό συναλλαγό σε διάφορα σημεία της έκθεσης, εγώ δεν έχω αντίρρηση αν όλοι συμφωνήσουμε, αλλά δεν θα ήθελα να μετατραπεί αυτό το σημείο σε επίμαχο. Γιατί αν δεν υπάρξει ευρεία συμφωνία υπέρ αυτών των τροπολογιών, θα ζητήσω και εδώ από τους συζητητές τους να τις αποσύρουν. Πρόκειται για, για τις τροπολογίες 36 και 138. Εγώ, όπω ξέρετε, είμαι υπέρ του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αν δημιουργηθεί εύκολα η συνένεση μεταξύ μα και μπορούμε να τι υπερψηφίσουμε, κανένα πρόβλημα. Αν όμω μετατραπεί αυτό σε έρηδα, σε μήλο έρηδα και σε σημείο αντιπαράθεση, προτιμώ να εμείνουμε στον αρχικό μα στόχο και να μην παρεκτραπούμε από την αρχική μα κατέθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες για την επανισορρόπηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και ιδιαίτερα της τροπολογίας μου για το κεφάλαιο 1, την δημιουργία λοιπόν ενός Ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών κατά κάποιο τρόπο, εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα εις βάθος, γιατί εγώ είχα υποβάλει αυτή την πρόταση ενός Ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών, αντίστοιχο παρόμοιο με αυτό το Αμερικανικού Υπουργείου, δηλαδή μιας αρχής που σε θέματα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής είναι ένας διαμεσολαβητής ή εταίρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως είναι στην Αμερική το Υπουργείο Οικονομικών απέναντι στη ΦΕΔ. Οι τροπολογίες του ΕΛΚ ναι, δεν αμφισβητούν αυτή την πρόταση, αλλά κάποιες τροπολογίες των πρασίνων και το συζήτησα μαζί τους προτείνουν αντικατάσταση αυτή της πρόταση για Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών με την πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο ή Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χρέους. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο φιλόδοξη αυτή η πρόταση σχέση με τη δική μου πρόταση. Και ούτε είναι και διφατική ε, ω προ την πρόταση του Ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών. Η δική σα ομάδα, κύριε Πρόεδρε, προτείνει διαγραφή αυτή τη πρόταση. Θα δούμε αν στην πορεία της συζήτησης μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση. Γιατί πιστεύω ότι αυτή θα ήταν μια χρήσιμη πρόοδος. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενημέρωση, την επικαιροποίηση, σε ό,τι αφορά τις μνήμες μας ε, για την αναθεώρηση της συνθήκης, Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια διατύπωση ώστε να λάβουμε υπόψη και τη φάση της αναθεώρησης για την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκα και στο βασικό ζήτημα του πρώτου κεφαλαίου. Τώρα για το δεύτερο κεφάλαιο είπα δύο λόγια για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. η πρόταση για την οποία αρχικά είχα ζητήσει και έκτακτη συνάντηση για να συζητήσουμε για το μέλλον ε, του G20 και ευελπιστώ ότι για το σημείο αυτό θα καταλήξουμε στη συμβαστική λύση γιατί το G20 δεν μπορεί να μετατραπεί σε Συμβούλιο Οικονομικής Ασφάλειας, αλλά ένα μεταρρυθμισμένο, ένα διαμορφωμένο G20, καλύτερα προσαρμοσμένο στην εκπροσώπηση των διαφόρων περιφερειακών ομάδων, θα μπορούσε να ενταχθεί στις προτάσεις μας. Ως προς το κεφάλαιο 3 τώρα. Εδώ έχουμε την πρόταση του πεδίου, την αναφορά του πεδίου ενός νέου ε, διεθνούς νομισματικού συστήματος. Έχουμε εδώ κάποιες τροπολογίες του, ε, του, των φιλελευθέρων. Θα πρέπει να δούμε και με το ΕΛΚ, για να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ό,τι αφορά την θέσπιση ενός ε, διεθνούς νομισματικού αποθεματικού. Τώρα το θέμα της συμπληρωματικότητας ό,τι αφορά τον, τις δαπάνες του, Ευρω... του κοινοτικού προϋπολογισμού και τις δαπάνες των εθνικών προϋπολογισμών ώστε να αυξήσουμε το επίπεδο των επενδύσεων, το ποσοστό των επενδύσεων και το ύψος των επενδύσεων στο μέλλον και για το σημείο αυτό θα χρειαστούμε κάποιες διευκρινήσεις για τη θέση του ΕΛΚ. Σε ό,τι αφορά τα σημαντικά για τις διαπραγματεύσεις σημεία. Στο κεφάλαιο 4 έχουμε το θέμα της παραγράφου 41 για την φορολογική εναρμόνιση και ιδιαίτερα για την ενιαία βάση του εταιρικού φόρου 3 CTB α6 στα γαλλικά. Για το σημείο αυτό υπάρχουν ενδιαφέρουσες τροπολογίες, μία των φιλελευθέρων που ξεφεύγει λίγο από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι προαιρετική και μια άλλη πρόταση που δίνει μια ψαλίδα ποσοστών. Υπάρχει και μια τροπολογία του ΕΛΚ σχετικά που προτείνει την αντικατάσταση της εναρμόνισης από το συντονισμό. Βέβαια δεν είναι τόσο φιλόδοξη η πρόταση αυτή. Γι' αυτό και δεν με βρίσκει ιδιαίτερα ενθουσιώδη. Ένα σημείο που με απογοητεύει αφορά την παράγραφο 43. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των διαρθρωτικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις ε, δημοσιονομικές στρατηγικές των κρατών μελών. Και εκεί θα πρέπει να φροντίσουμε να βρούμε μία διατύπωση συμβαστική, αλλά αξίζει να μπούμε στον κόπο. Σε ό,τι αφορά τις ε, δημόσιες επενδύσεις για την εκπαίδευση, και στα πλαίσια και του Συμφώνου Σταθερότητας, η δική πολιτική ομάδα είναι κατά και από ό,τι ξέρω το ΕΛΚ θα πρέπει και αυτό να διευκρινίσει τη θέση του. Αυτά για το, κεφάλαιο 4. Περνάμε στο κεφάλαιο 5. Η πρώτη παραγραφά όσο αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πολλέ τροπολογίε ζητούν την διαγραφή αυτή τη παραγράφου. Είναι μεμονωμένες όμως, δεν καλύπτονται από την υπογραφή των αντίστοιχων συντονιστών. Δεν είναι και πολύ χρήσιμες. Έχουμε όμως και μια τροπολογία του ΕΛΚ, το 428, που φαίνεται ενδιαφέρουσα. Το ίδιο ισχύει και για την παράγραφο 52, τη σχετική με την κοινοτική μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για την οικονομική διακυβέρνηση. Παράγραφος 55 αφορά το μέγεθος των διαφόρων δομών που εμπλέκονται στην, στην κεφαλαία αγορά και τη διαχωρισμό μεταξύ των ε, ταμιευτηρίων και των ε, επενδυτικών τραπεζών. Μερικοί ζήτησαν διαγραφή αυτής της παραγράφου. Το ίδιο ζητά και η τροπολογία 465 του ΕΛΚ που προτείνει διαγραφή αυτή τη σημεία. Νομίζω ότι αποτελεί τμήμα τη ε, γενική συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση. Δεν προεξοφλώ την έκβαση τη συζήτηση αυτή, αλλά η συμπεριφορά των τραπεζών από την κρίση και μετά νομίζω ότι μα δημιουργεί αυτόν τον προβληματισμό. Παράγραφος 57 αφορά την ε, ενίσχυση του κοινοτικού προϋπολογισμού χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένη συγκεκριμένο ποσοστό, μια ψαλίδα μεταξύ 5 έως 10% του ΑΕΠ μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν τροπολογίες για το θέμα αυτό που είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Έχουμε και μια τροπολογία του κυρίου Νταφ που δεν πάτησε πόδι στην Επιτροπή, στην δράση Επιτροπή Κρίσης, αλλά προτείνει τη μείωση στο 2,5% αυτή την ψαλίδα. Δεν τη λαμβάνω υπόψη, γιατί δεν νομίζω ότι μια τέτοια τροπολογία ανταποκρίνεται στις εργασίες της Επιτροπής μας. Το ΕΛΚ προτείνει διαγραφή αυτής της ψαλίδας προτείνει απλώς να αναφέρουμε γενικά μια φιλόδοξη αύξηση του κοινωτικού προϋπολογισμού. Με απογοήτευση σχετική τροπολογία του ΕΚ, του ΕΛΚ, γιατί άλλο να λέμε ότι θέλουμε φιλόδοξο προϋπολογισμό και άλλο να λέμε ότι μακροπρόθεσμα θέλουμε να φτάσουμε σε 5-10% του ΑΕΠ του ΑΕΠ. Καλύτερα να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Γι' αυτό προτιμώ να έχουμε αυτό το φάσμα, την ψαλίδα μεταξύ 5 και 10 και όχι απλώ τη διατύπωση φιλόδοξη, φιλόδοξος προπολογισμό. Σε ό,τι αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα δεν έχω πρόβλημα. Για την παράγραφο 59 και τις απαραίτητες ε, μελλοντικές αλλαγές για τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Έχουμε εδώ και κάποιες αντιφατικές τροπολογίες, ακόμη και από τις ίδιες ομάδες. Έχουμε αντιφατικές τροπολογίες των φιλελευθέρων, για παράδειγμα. Θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά. Ιδιαίτερη ικανοποίηση για την παράγραφο 61. Όλοι συμφωνούμε ότι η επόμενη θεώρηση συνθήκης θα πρέπει να γίνει με μια συνέλευση. Και μια μικρή έκπληξη με την παράγραφο 62, για την οποία έχουμε δύο τροπολογίες, μία του κυρίου Σμιτ και μία του κυρίου Νταφ, που θεωρούν ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να βαδίζουμε προς μια ενισχυμένη συνεργασία. Ενώ η αρχική διατύπωση, από ό,τι θα θυμάστε, προέβλεπε αν δεν καταφέρουμε να ενισχύσουμε την Ευρωζώνη, καλό θα ήταν να οδεύσουμε προς μια ενισχυμένη συνεργασία, αλλά όχι οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση. Δεν είμαι και πολύ θερμή για τις τροπολογίες αυτές. Γιατί κατά τη γνώμη μου δεν αντικατοπτρίζουν το πνεύμα το... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που με επιτρέψετε να μακρηγορήσω προκειμένου να κάνουμε την εισαγωγή αυτή τη συζήτηση που θα είναι και βάση για τι ε, αυριανέ συμβαστικέ λύσει. Ε, Σε ευχαριστώ το Είναι διεξοδική η παρουσίαση. Βλέπουμε ότι μελέτησε πολύ καλά όλες τι τροπολογίε και νομίζω ότι παρά το μεγάλο αριθμό των τροπολογιών έχουμε αυτή τη φορά τουλάχιστον περισσότερες πιθανότητε, από ό,τι την προηγούμενη να καταλήξουμε σύντομα σε μια καλή συμβαστική απόφαση. Πριν δώσω λόγο στου προσώπου ε, των ομάδων, θέλω να πω τα εξή ότι ήταν νωρίτερα την κυρία Στάρκεβιτσούτε, που ήταν ε, και μέλο τη Επιτροπή των Οικονομικών στην προηγούμενη θητεία. Ήταν σε μια συνεδρίαση παλαιών μελών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας με τον Πατ Κόξ. Και αυτό δεν είναι τώρα. Και τώρα θα ήθελα να συγχαρώ και την κυρία Χίμπνερ η οποία βραβεύτηκε με το βραβείο του αυτοκράτορος Μαξιμιλιανού για το έργο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια. Την Κυριακή της επανεμήθηκε. Και τώρα καλό του εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Τον κύριο Μπένσον καταρχάς από τη Δανία εκ μέρους του ΕΛΚ ο οποίος θα πρέπει να αποχωρήσει κάπου στις 4. Γι' αυτό το δίνουμε πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σχολιάσω. Να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Μπερές για τις προσπάθειές της μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία στο διαδίκτυο για τις εργασίες της Επιτροπής που είχα τη δυνατότητα να δω μέχρι τώρα μας δείχνουν τι απόσταση έχουμε διανύσει. Η έκθεση αυτή καλείται να είναι μια σοβαρή συνεισφορά για την παρούσα και μελλοντική συζήτηση για τη χρηματοπιστωτική κρίση και η συζήτηση αυτή θα κρατήσει αρκετό καιρό ακόμα. Σχετικά με τις τροπολογίες εμείς εκπροσωπούμε με δημοκρατικό τρόπο τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν είμαστε τίποτα περισσότερο. Η δημοκρατία είναι μια δύσκολη προσπάθεια την οποία όλοι πρέπει να επιχειρήσουμε. Μαζί με τον Χέρκμαρκ έχω προτείνει αρκετές τροπολογίες στο τελικό κείμενο. Δεν θα μιλήσω ε, εκ μέρους των υπολείπων που έχουν καταθέσει τις τροπολογίες, αλλά θα ήθελα να έχω στο τέλος μια έκθεση η οποία να είναι αναγνώσιμη. Μια έκθεση η οποία να ανοίγει δρόμους, η οποία όμως ταυτόχρονα να είναι αντιπροσωπευτική με αντιπροσωπευτικό τρόπο, εννοώ, την πραγματικότητα. Όχι υποχρεωτικά την αναζήτηση του χαμηλότερου κοινού παρανομαστή. Δύο πράγματα πρέπει να αναζητούμε. Πρώτον, να δούμε ποιες είναι οι φιλοδοξίες των εκλογιών μας. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε οι δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι Δεν είμαστε ούτε κυβερνητική η μη κυβερνητική οργάνωση, ούτε υπάλληλοι της Επιτροπής. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι νομοθετικός χώρος συζήτησης. Δεν είναι κάτι το οποίο θα καλύψει με νομοθετικό τρόπο τα θέματα των αυξήσεων του προϋπολογισμού κατά 5 ή με 10% με δεσμευτικό τρόπο. Κάτι το οποίο θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους πληθυσμούς της Ένωσης και τις μικρομεσαίες. Τέτοιες προτάσεις εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα προασπιστώ. Η χρηματοπιστωτική κρίση είναι αποτέλεσμα μιας μη ανεκτής πλέον δημόσιας δαπάνης και υψηλού δημοσίου ελλείμματος. Η λύση λοιπόν είναι να μειώσουμε το δημόσιο χρέος και να επιτρέψουμε την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Θα συμφωνήσετε μαζί μου κυρία Μπερές ότι για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή στους συμπολίτε μας όχι μόνο τις δικές μας ο καθένας τροπολογίες όχι μόνο αυτές τις οποίες συμφωνούμε πολιτικά, πρέπει να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε το πακέτο στο σύνολό του. Ελπίζω κάτι τέτοιο να είναι εφικτό όταν καταλήξουμε στην τελική ψηφοφορία. Κοφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ Προκαταρτικά θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις σχετικά με την μέθοδο εργασίας μας. Είναι προφανές ότι κάθε ένας από εμά εκπροσωπεί τους πολίτες που τον έφεραν εδώ. Σε κανέναν δεν μπορούμε να εμποδίσουμε να καταθέσει με τροπολογίες τις παρατηρήσεις του ή τα αιτήματα τροποποίησης στο υποσυζήτηση κείμενο. Αυτό είναι και η δημοκρατία. Η δημοκρατία όμως έχει και κανόνες και όχι μόνο συμβάσεις. Όταν παίρνουμε αποφάσεις, τις αποφάσεις αυτές πρέπει να τις σεβόμαστε. Εμείς αποφασίσαμε στις προηγούμενες συναντήσεις ότι οι συντονιστές θα έπαιζαν ένα ρόλο πολύ συγκεκριμένο. Έναν ρόλο συζήτησης στο εσωτερικό κάθε πολιτικής οικογένειας των τροπολογιών με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μειώσουμε τον αριθμό τους και να διευκολύνουμε τις καταληκτικές προσπάθειες του συνόλου της Επιτροπής μας και ιδιαίτερα της ηγήτριας. Παρατηρώ ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε σεβαστό. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους. Ε, με ένα σοσιαλιστής βουλευτής ε, κατέθεσε μια τροπολογία εκτός ελέγχου των συντονιστών θα τον εντοπίσουμε και θα τον τιμωρήσουμε αυστηρότατα, λέει ο εισηγητής, ο κύριος Κοφεράτη. Εν πάση περιπτώσει, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να κρατήσουμε μια τέτοια στάση απέναντι στις προσωπικές πρωτοβουλίες. Αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω ότι η προσπάθεια την οποία κάναμε εμείς σαν ομάδα δεν ακολουθήθηκε από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Το θέμα δεν είναι να αφήσουμε στην ιστορία ίχνη κυρωτικών πρακτικών ή γενικά αντιδράσεων σε μη ελεγχόμενες ενέργειες. Εν πάση περιπτώσει δραματοποιώ λίγο τα πράγματα, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Τίθεται ένα θέμα ουσίας εδώ. Όταν μετά από μια μακρά συζήτηση καταλήγουμε σε μια μέθοδο, καλό θα ήταν να την εφαρμόζετε τη μέθοδο αυτή. Έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, και εδώ είναι ένα επιπλέον δημοκρατικό κεκτημένο που δεν αμφισβητώ. Αλλά αυτές οι αλλαγές θέσεων νομίζω θίγουν την πολιτική μας οντότητα. Καταθέσεις τροπολογιών από συναδέλφων που ποτέ δεν καταδέχτηκαν να πατήσουν το πόδι τους στις συνεδριάσεις μας. Θεμητό είναι να το κάνουν νομικά. Πολιτικά όμως έχω την αίσθηση ότι η συμπεριφορά αυτή δεν είναι καλή. Εάν η συμμετοχή έχει κάποιο νόημα σε αυτή την περίπτωση, η συμμετοχή θα πρέπει να μην περιθωριοποιείται. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν με συγκεκριμένο τρόπο τώρα εξελιχθεί. Εγώ εξέφρασα τα παράπονά μου και ίσως να επανέλθω αργότερα σε αυτά. Μία παρατήρηση γενικού τύπου θα έλεγα στην περιγραφή την οποία η Περβάνς Μπερές ήδη έκανε με μεγάλη ακρίβεια θα έλεγα και επί της ουσίας. Επανειλημμένα έχουμε πει και είναι κάτι το οποίο πιστεύουν όλες οι πολιτικές οικογένειες με κάποιες λίγες εν πάση περιπτώσει εξαιρέσεις και αυτό φαίνεται από τις τροπολογίες ότι σε αυτή την κρίση εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε προωθώντας εκ νέου την εικόνα της Ευρώπης. Μια τέτοια κρίση αφορά φυσικά την Ευρώπη, εκδηλώθηκε στην Ευρώπη, λόγω ακριβώς των στρεβλώσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες και στο εσωτερικό των χωρών, αλλά έχει και χρηματοπιστωτική προέλευση. Και δεν είναι μόνο το έλλειμμα των κρατών που αποτελούν την Ευρώπη. Είναι, θα έλεγα, μία προσπάθεια η οποία α, πρώτα χτύπησε την οικονομία τον είπα και λόγω της παγκοσμιοποίησης έφτασε στην Ευρώπη και χτύπησε τα αδύναμα σκέλη θα έλεγα του χρηματοπιστωτικού και πιστωτικού ευρωπαϊκού συστήματος με άμεσες επιπτώσεις στα οικονομικά συστήματα των διαφόρων χωρών, ιδιαίτερα των πιο εύθραστων χωρών, αυτών που έχουν τα υψηλότερα ελλείμματα και που υπέφεραν περισσότερο. Όμως η λύση βρίσκεται στην ανάκαμψη της Ευρώπης Θα πρέπει λοιπόν, και το κάνω εγώ πρώτος αυτό, να προσπαθήσουμε να δούμε ποιο είναι το πολιτικό ε, μήνυμα που θα στείλουμε εμείς στη μέση της κοινοβουλευτικής μας εντολής. Όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε, οι συμβιβασμοί στους οποίους θα πρέπει να καταλήξουμε, θα πρέπει να έχουν σαν στόχο την ενίσχυση της Ευρώπης και τον εντοπισμό μιας πορείας μέσα από την οποία θα αυξηθεί και θα βελτιωθεί και δεν θα αποδυναμωθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αν απαντάμε σε οξυμένα κοινωνικά προβλήματα με την ιδέα της υπαναχώρησης ή της επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής διάστασης, τότε σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε κάνει ένα σοβαρότατο λάθος. Για μένα το κέντρο της τελικής μας πρότασης αυτό θα πρέπει να είναι. Αλλιώς δεν θα έχει χρησιμότητα η προσπάθειά μας. Αν απέναντι σε μια κρίση, μια ομάδα χωρών κατά περίπτωση βρίσκει λύσεις και αρνείται να προχωρήσει από κοινού προς τα εμπρός, αποδεχόμενη ε, την υπαναχώρηση και την επιστροφή στο παρελθόν σαν αναπόφευκτη, τότε είναι προφανές ότι μια τέτοια λογική εγώ δεν θα μπορέσω να την αποδεχθώ. Δεν υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις και τέτοια όρια. Στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί βέβαια υπάρχουν κάποιες τάσεις να προχωρήσουμε με μια Ευρώπη πιο συνεκτική, προς μια Ευρώπη πιο συνεκτική, μια Ευρώπη με ρόλους πιο ευρωπαϊκούς και λιγότερο εθνικούς. Και υπάρχουν αιτήματα για διάφορους τομείς όπως ο χρηματοπιστωτικός και ο τραπεζικός έτσι ώστε να εκχωρηθούν ορισμένες αρμοδιότητες ε, των οργανισμών αυτών, των χώρων αυτών προς τις νέες ευρωπαϊκές ε, οργανώσεις. Λοιπόν, τέτοιες ιδέες τις έχουμε κυκλοφορήσει. Τις ιδέες της ενίσχυσης της Ευρώπης. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτές τις ιδέες. Ελπίζω όλοι θα μας βοηθήσουν οι ιδέες αυτές, θα βοηθηθούμε από το να καταλήξουμε στις επιθυμητές ε, συμβιβαστικές λύσεις μένοντας πάντα πιστή σε αυτή τη βασική ιδέα εκκίνησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοφεράτη. Πριν να δώσω το λόγο στον επόμενο συνάδελφο, θα μου επιτρέψετε ίσω μια σύντομη απάντηση στον κύριο Μπέλτσεν, τον συνάδελφο που θα πρέπει να αποχωρήσει σχετικά σύντομα, μια και είπε ότι δεν είναι νομοποιημένη η Επιτροπή μα να συζητά θέματα των ιδίων πόρων, του προπολογισμού και Έχετε δίκιο ότι δεν μπορούμε να λαμβάνουμε απόφαση εδώ, γιατί δεν είμαστε νομοθετικό να νομοθετικών τον επιτροπή. Πλην όμω, ανεξαρτήτως το τι στάση τηρούν σε ορισμένε προτάσει, σε ορισμένε πολιτικέ ομάδε, έχουμε την αρμοδιότητα να διατυπώνουμε προτάσει για το μέσο πρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, όπως θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο. Και έχουμε δει επίσης πόσο μεγάλη σημασία έχει να ενημερώνεται και η κοινή γνώμη για το θέμα αυτό. Είδαμε στις τελευταίες εκλογές, σε παραδείγματι της Φινλανδίας, το 20% των ευρωσκεπτικιστών. Άρα ο πολίτης δεν είναι αρκετά ενήμερος σε ορισμένα ε, θέματα ευρωπαϊκά στις ε, χώρες μέλη. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα είναι καλό να ενημερώνεται περισσότερο, να ευαισθητοποιείται και όπως υπόθηκε και νωρίτερα, αν θέλουμε στο μέλλον να εμβαθύνουμε ε, στην ολοκλήρωση την ευρωπαϊκή στο μέλλον, καλό θα ήταν να κερδίσουμε περισσότερο τον πολίτη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να... ότι αυτό που λέτε δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να απόσχουμε κάποιες τοποθέτησεις ψηφοφορία μέσα στην Επιτροπή μας, αλλά ότι θα πρέπει να διατυπώσουμε τις θέσεις μας και αντίστοιχα να τις κοινοποιήσουμε, να τις νοσιοποιήσουμε και στην κοινή γνώμη. Και μια ακόμη παρατήρηση προς την Περβάνς για τις ε, τροπολογίες από τη δική μας πλευρά και με ορισμένου συγκεκριμένου συναδέλφων. Όπως είπα, είχαμε την ε, προεκλογική εκστρατεία στη Φιλανδία. Κάποιοι κατέθεσαν ε, ε, με το δικό τους όνομα την μία ή την άλλη τροπολογία, ενδεχομένως σκοπεύοντας να την παρουσιάσουν σε ορισμένα, υπό συγκεκριμένες συνθήκες στην προεκλογική εκστρατεία στη Φιλανδία. Ε, ο δε Άντριου Νταφ επικαλούμενος τον κανονισμό. Θέλησε να καταθέσει την τροπολογία. Εγώ του εξήγησα ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό, αλλά επέμεινε. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα σας πω ένα μυστικό και παρακαλώ να μην το πάρει το ποτάμι. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις απόψεων στην, στην ε, ομάδα των φιλελευθερών. Έχουμε διαφορετικές θέσεις από εδώ και από εκεί. Και έχουμε φερειπίν δύο συντονιστέ. Άρα δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τις μεθόδους που μας συνιστά ο Ιταλός συνάδελφο, γιατί αυτό θα σήμαινε 84 διαφορετικές πολιτικές ομάδες των φιλελευθέρων, δηλαδή 84 μέλη. Έτσι έχει η κατάσταση. Γι' αυτό και δεν μπορούμε. Και κύριε Κλέντ, δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε καν να, προσπαθ... να εμποδίσουμε τους συναδέλφους στη διατύπωση κάποιων θέσεων εδώ μέσα στην Επιτροπή αυτή. Εγώ νομίζω ότι συγκαταλέγομαι στους μάλλον φιλελευθέρους. Κάποιοι ίσως με θεωρούν δε και μάλιστα φιλελεύθερο. Αλλά για να απαντήσω στον δανό συνάδελφο Μπορεί να σας φαίνεται κάπως προκλητική η έκθεση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να τη θεωρήσει κανείς και όραμα. Ένα όραμα το οποίο εσείς μπορεί να μην συμμερίζεστε, αλλά πάντως είναι όραμα. Πιο συγκεκριμένο σε ορισμένους τομείς, λιγότερο συγκεκριμένο σε, κάποιο άλλους, σε κάποιους άλλους. Και αυτό είναι η προσωπική μου γνώμη που θα πω. Ότι δηλαδή, όπω είχαμε αποφασίσει στην ΕΚΟΝ, το Κοινοβούλιο και βέβαια και το Συμβούλιο κτλ., είχαμε 18 μήνε μπροστά μα. Λοιπόν, εάν πριν από 18 μήνε έλεγε κανεί, Α, θα σα κάνω την πρόβλεψη ότι αυτό και αυτό θα συμβούν στην Ευρώπη, θα μα λέγανε είσαστε τρελοί. Και όμω συνέβησαν αυτά τα πράγματα και έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Κάποιε λοιπόν εκ των προτάσεων τη κυρία Μπερέ, ίσω στην αρχή να ήταν στον τομέα του οραματισμού μάλλον. Τώρα όμως είναι νομοθετήματα, είναι ήδη νομοθετημένες διδάξεις. Δεν είμαι λοιπόν τόσο ματαιόδοξο ώστε να ισχυριστώ ότι δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί δυστυχώ έχει αποδειχθεί ότι η ιστορία μπορεί να προχωρήσει με του ρυθμού. Αλλά κύριε Μπερέ, μου θυμίσατε μερικέ φορέ τη δασκάλα μου στο σχολείο που ήταν αυστηρή και με το χάρακα μου έλεγε παραείσαι εσύ άτακτο παιδί και με κοπάναγε. Εν πάση περιπτώσει θα το αντέξω και αυτό. Ξέρω ότι εάν με, κολα... με τιμωρήσατε ήσασταν ε, καλοπροαίρετοι. Επίσης θέλω να σας συστήσω να παρακολουθήσετε το Free City όπου έχουμε τέσσερι διαφορετικέ ε, απόψει των ε, φιλελευθέρων. Να σα πω. Στα ευρωομόλογα, Φερρυπίν. Ή στην οικονομική διακυβέρνηση. Εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ίσως όχι όλοι, Και πρέπει να πω ότι ύστερα από 8 μηνών ε, αντιπαραθέσεις με ξαφνιάζει κιόλας το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε στην ομάδα της Οικονομικής Επιτροπής των Φιλελευθέρων. Εντυπωσιακό. Για το Υπουργείο Οικονομικών, ναι, διαφωνούμε με ένα, αλλά η διατύπωση είναι τέτοια που ίσως να την δεχτείτε την πρότασή μας. Προϋπολογισμός. Ίσως είναι πιο δύσκολο θέμα γιατί βέβαια θα πρέπει να ακολουθήσουμε όρους συνεπείς με αυτά τα οποία λέει και η ΣΟΥΡ. Επίσης κάναμε με την παρουσία και της Ουγγρικής Προεδρίας ε, στη Στοκχόλμ μια συνεδρίαση. Είδαμε ταυτόχρονα και τον Ολλανδό ε, πρεσβευτή στη συνεδρίαση αυτή και βέβαια ξέρετε όλοι τι λένε οι Βρετανοί, οι Σουηδοί και οι Ολλανδοί ε, για το θέμα αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Το Κοινοβούλιο πρέπει στα θέματα αυτά να δράσει με πολύ μεγάλη σύνεση. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να φωνάζουμε δεξιά και αριστερά, θα έχουμε και άλλα λεφτά. Γιατί ενδέχεται να χάσουμε και αυτά που έχουμε στη διάθεσή μα. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε εμεί το μόνο θεσμικό όργανο, το μόνο πολιτικό θεσμικό όργανο στην Ευρώπη που δεν μιλάει για λιτότητα. Φορολογία. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα πρέπει να διατυπώσετε συμβαστικές προτάσεις, συμβαστικές τροπολογίες. Θα διαπιστώσατε ότι και εκεί διαφοροποιούμαστε. Μάλλον εκφράζουμε διαφορετικές απόψεις. Ε, αλλά πιστεύω τελικά θα σας ακολουθήσουμε. Εάν μπορέσουμε να, αν μπορέσαμε μάλλον την προηγούμενη φορά να καταλήξουμε σε συμβαστικέ προτάσει, θα τα καταφέρουμε και τώρα. Μετά μου λέτε για την παράγραφο 62 και τις δύο τροπολογίε που έχουμε σε αυτήν. Είναι τόσο πια απίθανο. Μου το δεχτείτε. Εσείς λέτε πιστεύει ότι μπορεί να εμείς λέμε ότι, ε, ότι αν αυτό δεν συμβεί και εμείς λέμε ότι σε κάθε περίπτωση. Πιστεύει ότι σε κάθε περίπτωση. Είναι πια τόσο τεράστια η διαφορά. Για δε τον Άντρου Νταφ καταλήγω λέγοντας ότι δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ότι δεν είναι καλός Ευρωπαίος. Ε, ευχαριστώ πιέτικα Κάινεν τώρα. Κυρία πιέτικα Κάινεν, η οποία από ό,τι κατάλαβα θα παρουσιάσει την επίσημη θέση του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Uh, και σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Μπορώ να το ομολογήσω. Είναι από τις κακές συνήθειες που έχω. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν ε, χτυπάω μικρά ζώα. Ήδη άκουσα την ενημέρωση της συγκεκριτής κυρίας Μπέρες και τα σχόλιά της για τις τροπολογίες και θα προσπαθήσω να τη σχολιάσω και να προσθέσω και κάποιες σκέψεις. Εμείς στο ΕΛΚ θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και προσπαθούμε να προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τον αριθμό των τροπολογιών επιμένοντας τα σημεία που θεωρούμε ότι θα συγκεντρωθεί συνένεση για συμβαστική λύση και προσπαθούμε να είμαστε και όσο πιο φιλόδοξοι πολιτικοί γίνεται στην ομάδα μας. Ευχαριστούμε την εισηγητριά μας για την καλή προεργασία που έκανε, για όλες τις προσπάθειές της στην Επιτροπή που ήταν πολύ επικοδομητικές και μας δημιουργήσαν και μια πολύ στέρη βάση για την περαιτέρω ε, συζήτηση μεταξύ μας. Νομίζω ότι οι τροπολογίες μας χαρακτηρίζονται από φιλοδοξία και για την οικονομική διακυβέρνηση, για το Υπουργείο Οικονομικών και τα επόμενα βήματα. Σε ό,τι αφορά το προπολογισμό, αν θα λέμε φιλόδοξο προπολογισμό, θα πρέπει να αναφέρουμε και μια ψαλίδα με ποσοστά. Δεν νομίζω ότι είμαστε στο ΕΛΚΑ διάλακτοι, τελείω αδιάλακτοι για το θέμα αυτό, αλλά θα πρέπει να λάβουμε ορισμένα στοιχεία υπόψη. Φυσικά δίστανται οι απόψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε να ευθυγραμμιστούμε με την Επιτροπή ΣΟΥΡ και με την αντίστοιχη έκθεση και να είμαστε συνεπείς ε, και συμβατοί με τις δικές τους προτάσεις. για να μην δημιουργηθεί διχασμός μεταξύ των δύο επιτροπών. Και να έχουμε υπόψη το στόχο και να δούμε τι θα μας εξυπηρετήσει περισσότερο. Να μιλούμε για φιλόδοξο προϋπολογισμό ή να αναφέρουμε συγκεκριμένα ποσοστά. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση, την εναρμόνιση, το συντονισμό μάλλον ή την εναρμόνιση. Και αυτό το θέμα το συζητήσαμε πολύ. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, θέλουμε να γίνουν κάποια επικοδομητικά βήματα στην Επιτροπή μας και να θέσουμε το ζήτημα των ιδιών πόρων και έχουμε και το θέμα του FTT παρόλο που ξέρουμε ότι υπάρχουν διστάμενες απόψεις και προσπαθούμε να συμμετέχουμε όσο πιο ε, επικοδομητικά γίνεται στη συζήτηση και σε ό,τι αφορά τα ευρωομόλογα επίσης. σε ό,τι αφορά τα θέματα τα επενδυτικά, τα τραπεζικά, δεν είμαστε και το διαχωρισμό των τραπεζών, δεν είμαστε απόλυτα αρνητικοί, αλλά διαρωτόμαστε πόσο απαιτητικοί θα πρέπει να είμαστε στο σημείο αυτό. Τώρα, για τον αριθμό των τροπολογιών και το ποιος τις κατέθεσε, εμείς είμαστε πολύ ενεκτική ομάδα και δίνουμε έμφαση στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε ένα χάρακα ή να επιβάλλουμε κυρώσει και τιμωρίε. Ο καθένας υποβάλλει κατά το δοκούν τις τροπολογίε που θεωρεί χρήσιμες. Πάντως συμφωνήσαμε και με μια διαδικασία Γι' αυτό και η στεπτική πλειοψηφία της ομάδας μας θα υποστηρίξει αυτή τη γραμμή της ομάδας και στόχος μας είναι να καταλήξουμε στο μέτρο του δυνατού σε μια ισχυρή έκθεση που θα συγκεντρώνει ευρύτατη συνένεση έως και ομοφωνία γίνεται. Βέβαια υπάρχουν και μεμονωμένοι βουλευτές που έχουν το δικαίωμα να ταχθούν υπέρ των δικών τους τροπολογιών. Ευχαριστούμε Σερμπά. Κυρία Χιμπνερ. Ευχαριστώ. Να πω ότι είχα και εγώ τη δυνατότητα να συνεισφέρω στην έκθεση Βερές με ένα κείμενο εργασίας για τη χρηματοδότηση της μελλοντική ανάπτυξης στην Ευρώπη. Και είμαι ευγνώμων γιατί περισσότερες από τις ανησυχίες μου έχουν γίνει δεκτές στην έκθεση της Βερές. Και είμαι σε καλή παρέα γιατί βλέπω και τις προτάσεις τις οποίες καταθέτει η Μπερές μαζί με τρεις επιπλέον τροπολογίες που συνδέονται με το ότι για μας η Ευρώπη δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να διαβυνθεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τις αναπτυξιακές δυνατότητες και τις μεταρρυθμίσεις. Θεωρώ επίσης ότι έχει αρκετά μεγάλη σημασία εδώ να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο για να υπάρξουν αυξήσεις στις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας. Ελπίζω επίσης ότι θα μπορέσουμε στα πλαίσια των συμβιβαστικών τροπολογιών να βάλουμε και την ιδέα της στήριξης της ανάπτυξης των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων για την, μελλοντική της, ε, για την ανάπτυξη της, ε, τη, τη μελλοντική ανάπτυξη και την ε, αλλαγή και μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ. Όντως, η έκθεση αυτή απαρτίζεται από 63 σημεία, είναι την αιτιολογική έκθεση. Γι' αυτό και συγκέντρωσε τόσες τροπολογίες. Είναι λογικό σε μια τόσο περίπλοκη έκθεση και δεν μας εκπλήσει ο αριθμός 522. Πάντως ήταν ε, καλό το έργο της συγκήτριας, πολύ πετυχημένο και κατάφερε να παρουσιάσει ένα συγκροτημένο σχέδιο και να διαρθρώσει πολύ καλά την έκθεσή της. Εγώ ασχολήθηκα με το συντονισμό των εργασιών στη σοσιαλιστική ομάδα και όπως θα είδατε κατέθεσα δύο μόνο τροπολογίες με δική μου υπογραφή μόνο. Οι υπόλοιπε ήταν οι, οι γενικές τροπολογίες της ομάδας με την υπογραφή του συντονιστή. Και μάλιστα για την πρώτη τροπολογία και ο συντονιστής και η συγγήτρια έδειξαν μεγάλη ανοχή και ελαστικότητα. Στην πρώτη τροπολογία αυτό που με προβλημάτισε είναι να δούμε ποια σχέση υπάρχει μεταξύ του εξωτερικού χρέους, του δημόσιου χρέους μάλλον και της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Και θέλουμε να έχουμε, καλ... έχουμε καλά... καλούς δημόσιους λογαριασμούς και εξηγήσεις των οικονομικών. Και μπορεί το θέμα αυτό των, ε, της κρίσης και του δημόσιου χρέους να φαίνονται ξεχωριστά, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια ισορροπία υπάρχει μεταξύ τους. Σε πολλές περιπτώσεις δεν αναγνωρίζεται ρητά η σχέση τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε όμως ε, κατηγορηματικά, γιατί μιλάμε για συστημικές καταστάσεις και το χρηματοπιστωτικό κλάδο, γι' αυτό και μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι και οι χώρες ε, έχουν συστημικό χαρακτήρα γιατί πραγματικά έχουν τεράστια σημασία για τους πολίτες χάρη στις, στα αγαθά που τους προσφέρουν και τις βιωτικές συνθήκες που παρέχουν. Αυτό το ζήτημα έθεσα με την πρώτη μου τροπολογία. Στη δεύτερη τροπολογία, μια και η Επιτροπή μας έγινε για την ε, χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, προσπάθησε στη δεύτερη τροπολογία να επισημάνω ένα θέμα που δεν έτυχε της δέουσας προσοχής της εργασίας μας ενώ είναι πολύ σημαντική γιατί αφορά την κοινωνική πτυχή της κρίσης που είναι, αναφέρεται και στον τίτλο της Επιτροπής μας. Και βέβαια η κοινωνική πολιτική φαίνεται να είναι ευθύνη του κάθε κράτους και να, είναι, να έχει πιο τομεακό χαρακτήρα. Αλλά το, πλαίσιο των, το μακροοικονομικό πλαίσιο των κοινωνικών πολιτικών και η ευρύτερη δημοσιονομική και οικονομική προσανατολισμή μας μπορούν να προσανατολίζουν και να συμβάλλουν στην κατεύθυνση που λαμβάνει μια κοινωνική πολιτική. Οπότε από αυτή την άποψη αναγνωρίζοντας ε, το θέμα της οικονομικής ανάκαμψης, της στρατηγικής 2020, ε, τα δημόσια οικονομικά και την προσπάθεια εξυγίαση των δημόσιων λογαριασμών είναι θέματα που αναφέρουμε στην έκθεση, αλλά όλα αυτά σε τελική ανάλυση δεν αρκούν. Γιατί δεν αρκούν οι υπάρχουσε πολιτικέ. Γιατί έχουμε και πάλι αβεβαιότητα και αδυναμίες στην Ευρώπη. Χρειάζεται και ένα επιπλέον στοιχείο, να συμπληρωθούν όλα αυτά ώστε να έχουν νόημα για τους πολίτες. Χρειαζόμαστε ένα κοινωνικό σύμφωνο αυτό το κοινωνικό σύμφωνο έχει τρεις σαφέστατε διαστάσεις. Καταρχήν θα πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα και είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα γενικότερο πλαίσιο και ραγδαία παγκοσμιοποίησης και αύξηση της ανταγωνιστικότητας από τις αναδυόμενες οικονομίες και τους νέους εταίρους θα πρέπει να επανεπιβεβαιώσει τις βάσεις της ανταγωνιστικότητάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως αυτό να το κάνει και με ένα κοινωνικό σύμφωνο. Αλλιώς θα υπονομευθούν ε, τα ίδια τα θεμέλια της ευημερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη διάσταση συνδυάζεται με ένα γενικότερο θέμα που είναι αυτό το, το φορολογικού βάρους. Το θέμα αυτό δεν είναι ίσονο σημασία, γιατί βλέπουμε πως ε, Έχουμε την έμεση φορολογία, τη φορολογία της εργασίας, που αποκτούν όλο και περισσότερη σημασία στους εθνικούς προϋπολογισμούς και έχουν ε, χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο και δημοσιονομικό σημαντικό αντίκτυπο. Έτσι φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι κάποιοι κλάδοι απολαμβάνουν ε, τα προνόμια της οικονομίας αλλά δεν ε, αναλαμβάνουν αντίστοιχα και τις υποχρεώσεις γιατί είχαμε αύξηση των εσόδων ορισμένων κλάδων, αλλά ελάχιστη συνεισφορά αυτών των κλάδων στην, ε, στις δημόσιες δαπάνες. Αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε στις μελλοντικές βάσεις ε, της ευημερίας μας. Ένα τρίτο ζήτημα που είναι συναφές με τα προηγούμενα αφορά την ενίσχυση, την επικαιροποίηση του του κράτους πρόνοιας ή της ευημερία. Μερικοί θεωρούν ότι αυτό, αυτή η κατάσταση της ευημερία και το κράτος πρόνοιας είναι η απάντηση που δόθηκε για να αντιμετωπιστούν κάποιες μόνιμες ανάγκες της υγείας, της παιδείας, ανάγκες αντιμετώπισης κινδύνων. Αυτές οι ανάγκες είναι πρωταρχικές. Δεν ε, καταργούνται αυτές οι ανάγκες. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μία στέρεη οργάνωση και ένα σύστημα στο μέλλον ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες και στο νέο πλαίσιο. Αυτά τα σημεία λοιπόν τα νέα επισήμανα στις τροπολογίες μου και νομίζω ότι είναι η τελευταία αυτή τροπολογία ούτως ή άλλως που εστιάζει την προσοχή μας σε κάποια άλλα σημεία και ίσως δεν τα αναλύσαμε πιο διεξοδικά γιατί ξεφεύγουν από τις αρμοδιότητές μας αλλά είναι θέματα που θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε και να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας στα πλαίσια που προχωρούμε στις εργασίες μας και καθορίζουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τρεις συνάδελφοι ακόμη αυτοί που είχαν ζητήσει το λόγο. Ρωτώ αν ακόμη θέλουν να, λάβουν, ε, να μιλήσουν. Η κυρία Ρόιτκοβα από το ΕΛΚ. Ρωτάω αν ακόμα επιμένετε. Ο κύριος Δημένιτσι. Κύριε Γκόνς, ναι. Όχι. Κύριος Δομένιτσι. Η κυρία Ρότκοβα. Έτσι και έτσι. Θέλετε το λόγο. Όχι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την κυρία Γκέντς. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη γιατί καθυστέρησα, αλλά έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό τροπολογιών δυστυχώς. Κάποιες από αυτές συγκλίνουν, κάποιες όμως δυστυχώς αποκλίνουν η μία από την άλλη. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις επί τη βάση συγκεκριμένων αρχών που προτείνουμε, εμβαθύνοντας και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ελπίζω να καταλήξουμε σε μία κοινή διατύπωση η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης σημαίνει εμβάθυνση πολιτικής συνεργασίας, οικονομικής συνεργασίας και έχει πολύ μεγάλη σημασία στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ολοκλήρωσης να υπάρχουν και οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των αναγκών αυτής της ε, ολοκλήρωσης. Βλέπουμε ότι σε διάφορους πολιτικούς τομείς προχωράμε. Κάποιοι από τους τομείς αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικοί για το ξεπέρασμα της κρίσης και αναφέρομαι στην εκπαίδευση, στο περιβάλλον, στη διαβίου κατάρτιση, στην παιδεία. Εκεί είναι ξεκάθαρες οι αναπτυξιακές μας αρχές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και τη στρατηγική του 2020 στα πλαίσια ακριβώς αυτού του τρόπου αντιμετώπισης των μελλοντικών προβλημάτων είναι επίσης οι πρωτοβουλίες flagship απαραίτητο να εξυπηρετηθούν σωστά και ταυτόχρονα να αποφύγουμε την περίοδο πριν από την στρατηγική της Λισαβόνας γιατί κάτι τέτοιο θα υπονομεύσει ουσιαστικά τις θετικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών. Ελπίζω και η κοινότητα ενέργειας της Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης να συμπεριληφθεί στην τελική πρόταση. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μείζωνα προβλήματα γύρω από το θέμα της ενέργειας. Είχα και ορισμένες τροπολογίες ετοιμάσει επίσης για να αποτρέψουμε την ανάπτυξη μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων που είναι σημαντικό κίνδυνος για την Ευρώπη στο μέλλον. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια κάποια διατύπωση εδώ η οποία να γίνεται αποδεκτή από όλους. Ελπίζω λοιπόν ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ. Και σύντομα τώρα, αν μου επιτρέπετε να πω και εγώ δύο λόγια. Ο Λεσμίτ, ο συντονιστή, νομίζω εξέθεσε όλα τα ουσιώδη ζητήματα. Απλώ ήθελα εγώ να αναφερθώ σε μία πτυχή. Και σε σχέση με αυτά που ο κύριο ήταν στην αρχή θα ήθελα να επισημάνω ότι θα είναι καθοριστική σημασία στο να προσδιοριστεί, το να διαμορφωθεί αυτή η έκθεση κατά τρόπο ώστε ο αναγνώστης που θα βρεθεί, θα την πάρει στα χέρια του, να μπορεί να αντιληφθεί, ακόμη και αν είναι ο κοινό πολίτη, πώς μπορεί να την αξιοποιήσει. Δηλαδή πώς πρακτικά προβλέπεται να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις να υπάρχουν ιδέες για πρακτικές εφαρμογές. Έχουμε μπροστά μα ένα φαινόμενο ευρωσκεπτικισμού σε πολλά κράτη ανωδικό και ως εκ τούτου θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει την έκθεση αυτή να την κάνουμε όχι για μα, όχι για αυτόν τον ε, γραφειοκρατικό κολοσσό που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρυξέλλες, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να θυμόμαστε πάντα ότι αυτήν την έκθεση τυπώνουμε γιατί έχουμε σαν κύριο μέλη μα ανάγκε και του προβληματισμού των πολιτών τη Ευρώπη και ότι θέλουμε να βοηθήσουμε να βελτιωθούν οι συνθήκε ζωή του με αυτήν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εκεί πρέπει να γίνει λίγο, λίγο περισσότερη δουλειά. Πολλά από τα αρχικά ε, σημεία της έκθεσης, από τις παραγράφους έκθεσης, αλλά και πολλές από τις τροπολογίες δεν ανταποκρίνονται σε αυτήν ε, την προϋπόθεση και γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να αναδιατυπωθούν κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε την έκθεση αυτή να την παρουσιάσουμε και θα έλεγα με θάρρος και πειθό να, και αυτοπεποίθηση να την παρουσιάσουμε στην κοινή γνώμη. Δεν είναι δηλαδή κάτι το αφηρημένο αυτή η πρόταση. Καλό θα είναι να καταλάβει ο πολίτης αυτό που λέμε στα αγγλικά what's in there for me, δηλαδή τι θα του προσφέρει στα επόμενα 5-10 χρόνια αυτή η έκθεση σε συγκεκριμένου όρου. Και νομίζω ότι θα πρέπει η Πεγός, ε, ίσω και με τη δική μα βοήθεια, να αναλογιστεί λίγο περισσότερο πώ θα μπορούσε να ενισχύσει το κείμενο υπ' αυτή την έννοια. Δίνω λοιπόν τώρα το λόγο στην Πεγός για κάποιε καταληκτικές παρατηρήσει με μία μόνο παρατήρηση ότι η προσοχή μα συνεδρίε είναι στι 23 του μηνό και είναι Δευτέρα. 23 του μηνό, οι συντονιστέ και οι σκιώδει ηγητέ, γιατί έχουμε και τετάρτη συνεδρίαση, για να συζητηθούν για άλλη μια φορά οι συμβαστικές ε, προτάσεις. 23 του μηνό Δευτέρα, επαναλαμβάνω, οι σκιώδει. Στις 25, δύο μέρε μετά, η Επιτροπή ε, στην Ολομέλειά τη, Και πιστεύω ότι στις 30 του μηνό θα μπορέσουμε να διεξαχάχουμε την ψηφοφορία μα Πεγόν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα επιβεβαιώσετε με mail στο σύνολο των μελών μας τις πληροφορίες που ακούσαμε, οι οποίες μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε τη χρήση του εναπομείνατος για τη διαπραγμάτευση χρόνου. Εδώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τους ε, συνεισηγητές και τους κοιόδης εισηγητές έτσι ώστε να τους αποστείλω μέχρι την Δευτέρα το απόγευμα μια άλλη πλέον βελτιωμένη πρόταση. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους οι οποίοι πήραν μέρος σε αυτήν την συζήτηση, σε αυτή τη φάση ακριβώς των εξελίξεων. Κύριε Πρόεδρε, εν πολλής έχετε ήδη απαντήσει στον συνάδελφο Μπέντσεν, ο οποίος δεν είναι πλέον μαζί μας. Κρίμα, ναι ξέρω είχε πει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να μιλήσω μαζί του σε διμερές επίπεδο, θα το επιδιώξω στο Στρασβούργο, είναι σημαντικό να μπορέσω να το απαντήσω. Και να επανέλθω επίσης και στο θέμα ε, του δημοσιονομικ... της δημοσιονομικής ψαλίδας εγώ θα έλθω σε επαφή με τους συναδέλφους που είναι μέλη της Επιτροπής μας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση η οποία ανακαλύπτει τις ανησυχίες τους. Να μου επιτρέψετε να σας θυμίσω όμως ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικούς ορίζοντες. Εμείς έχουμε ηθελημένα, εσκεμένα διαμορφώσει το χρονοδιάγραμμά μας σε σχέση και με τους άλλους συναδέλφους, γιατί και η προσπάθειά τους σταδιακά ακολουθεί τη δική μας αλλά ο δικός μας ορίζον δεν είναι ίσως, δεν, είναι, δεν ταυτίζεται με τις δημοσιονομικές πρόπτικες. Και ευχαριστώ τον Όλε Σμιτ, ο οποίο είπε ότι κάποιε από τι προτάσει οι οποίες έχουν κατατεθεί τον εκπλήσουν. Ε, ιδιαίτερα κάποιε από τι προτάσει τι οποίες έχω κάνει εδώ και κάποιο καιρό θα, ήταν, είχαν θεωρηθεί ιδιαίτερω πρωτοπόρε τολμηρέ. Παρ' όλα αυτά Λαμβάνοντας υπόψη την ένταση που έχει δημιουργηθεί από την κρίση έγιναν αντιληπτές ότι είναι ρεαλιστικές ε, τάχιστα. Σημερίζομαι λοιπόν την αίσθησή σας τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Παρ' όλα αυτά εξακολουθώ να είμαι πεπισμένη και νομίζω ότι πολλοί το πιστεύετε κι εσείς ότι το παρόν στάδιο εξέλιξης και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μακροπρόθεσμα υποστηρίξιμο. Ο Ζακ Ντελόρ μας το είχε πει όταν μας είχε επισκεφθεί τελευταία είπε ότι η κυρία Μπερές ε, είναι πολύ σημαντική, ε, συγγνώμη, πολύ φιλόδοξη και ότι σε αυτή τη φάση αυτό για το οποίο μιλάμε είναι η συνεργασία. Νομίζω ότι όπως έλεγε και ο Παντίας Κιώπα, νομίζω ότι πράγματι αυτό χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση αλλά έχω την αίσθηση ότι μέσω πρόθεσμα το ευρώ δεν θα επιβιώσει εάν δεν έχουμε ένα προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να επιτρέπει να θέσουμε σε λειτουργία αντικυκλικές πολιτικές. Να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα στοιχείο το οποίο και η Ελίζα Φερέρα υπογραμμίζει και το οποίο υιοθετώ πλήρως γιατί έχω την αίσθηση ότι πρέπει να μας προβληματίσει. Όταν είχε έρθει ο Παπανδρέου να μας συναντήσει στα πλαίσια της συνεδρίασης της Επιτροπής για την κρίση, είχε πει ότι λόγω των δεσμεύσεων τις οποίες απαιτεί από την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως να είχαμε μεγαλύτερο συμφέρον να πάμε στο Δέλτα Νιτάφ, γιατί τότε σε αυτή την περίπτωση αυτά που έχουμε ήδη κάνει θα τα αναγνώριζαν. Αν η Πορτογαλία πήγαινε στο Δέλτα Νιτάφα ε, σήμερα μόνο, ε, θα είχε δικαίωμα σε βοήθεια. Το θέμα δεν είναι αν θα δοθεί ή όχι η βοήθεια. Σήμερα, στα πλαίσια των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν λέω θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία δυνητικά ένα κράτος μέλος θα μπορούσε να αντιταχθεί σε αυτή την βοήθεια και να μην υπάρξει βοήθεια. Αυτή λοιπόν η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γι' αυτό λοιπόν μέσω πρόθεσμα έχω την αίσθηση ότι έχουμε ανάγκη από έναν πιο συνεκτικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ένα παρεμβατικό με δημόσιο βάρος προϋπολογισμό. Εκεί που συμφωνήσω με τον Όλε Σμίτ είναι ότι και εγώ δεν λέω ότι απαιτούνται περισσότερα χρήματα. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά πιστώσεων από τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μόνιμα ποσοστά κάθε φορά. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά όταν διατυπώσουμε την τελική συμβιβαστική πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον μιλάμε για με ένα σταθερό ποσοστό, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Και νομίζω ότι με τη λογική αυτή θα υπάρξει μια κάποια συμφωνία μεταξύ μας. Ευχαριστώ λοιπόν τον Σμιτ για τις παρατηρήσεις του. Είπε ότι η φιλελεύθερη ομάδα είναι τόσο φιλελεύθερη που έχει πολλές απόψεις. Ε, το γνωρίζω αυτό. Αυτό που μου είχε ξεφύγει είναι η αναφορά την οποία κάνατε στην φυσική σας αισιόδοξη πλευρά του χαρακτήρα. Και αυτό θα συνεχιστεί ελπίζω. Για την παράγραφο 62. Εδώ μου δίνετε την ευκαιρία να διευκρινίσω μια κάποια σύγχυση η οποία δημιουργήθηκε από τα πρώτα σχόλια. Μακράνε μου η ιδέα να θεωρώ ότι εσείς ή ο Νταφ δεν είστε πραγματικοί Ευρωπαίοι. Δεν εννοώ ποτέ κάτι τέτοιο. Η αίσθησή μου είναι, όπως είπε και ο προλαλής σας συνάδελφος, ότι το αν πούμε σήμερα ότι όπως και να έχουν τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στην βελτιωμένη ή ενισχυμένη συνεργασία είναι κάτι το οποίο θα προκαλέσει προβλήματα μεταξύ μας. Εγώ σαν Γαλλίδα σοσιαλίστρια είχα αλλάξει γνώμη. Εγώ παλιά ήμουνα υπέρ της ενισχυμένης συνεργασίας και του πρωτοπορία και του πρώτου κύκλου κτλ. Άλλαξα γνώμη όμω. Άλλαξα γνώμη γιατί ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εσωτερικό τη και προ τα έξω είναι να παραμένει ενιαία και ενωμένη. Αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι τα μέλη της ζώνης ευρώ σήμερα έχουν ιστορικές ευθύνες μπροστά τους, τι οποίες όμως θα πρέπει να αναλάβουμε ελπίζω με 27 χώρες. Αν δεν το πετύχουμε τότε θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο της ενισχυμένης συνεργασίας. Λοιπόν, πετικά είναι. Ευχαριστώ για το πνεύμα της ε, παρέμβασής σας που αντικατοπτρίζει την πλειοψηφία των μελών της πολιτικής σας ομάδας για τον προϋπολογισμό Απίνησα. δεν νομίζω ότι πρέπει να επανέλθω. Νομίζω ότι στη συμβιβαστική πρόταση θα βάλουμε ό,τι είναι χρήσιμο για την Επιτροπή μας, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και τις εργασίες των άλλων Επιτροπών. Για την 465, τροπολογία 465, υπάρχει πλήρης κατάργηση, πλήρης διαγραφή. Για μια στιγμή διακόπτει ομιλήτρια. Λοιπόν για την 465 κατάργηση όλου του τμήματος ε, στην αναφορά για τη διάκριση ανάμεσα στις, ε, στα ταμεία παρακαταθήκων και στις επενδυτικές τράπεζες. Γιατί όχι. Θα πρέπει να δούμε όμως εδώ τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι στην Ευρώπη δεν μπορούμε το θέμα αυτό να το θεωρούμε ταμπού. Ευχαριστώ και την Τανούτα για την αξιολόγηση τη θετική των εργασιών μου και για τις τροπολογίες της. Οι περισσότερες μπορεί να γίνουν δεκτές χωρίς καμία δυσκολία, ίσως όχι στην συγκεκριμένη θέση που προτείνεται, αλλά σε διαφορετικά σημεία του κειμένου, αλλά είναι τροπολογίες οι οποίες είναι πάντα χρήσιμες. Εγώ ανησυχώ λίγο γιατί από τη μία δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία έχουμε ήδη πει στην πρώτη έκθεση και από την άλλη θέλω να μην ε, μακρηγορήσουμε ιδιαίτερα εφόσον ε, επαναλαμβάνοντας αυτά τα οποία είπε ο Πρόεδρος πρέπει να είμαστε συνοπτικότεροι της πρώτης φοράς. Θα δούμε πώς θα το καταφέρουμε αυτό και εάν. Για τον Σάντσες. Είπε ότι αυτοκαταγγέλθηκε, είπε ότι εγώ είμαι ο σοσιαλιστής ο οποίος ε, δεν σεβάστηκα τον κανόνα της ομάδας Αποκαλύφθηκε λοιπόν μόνος του. Θα δω τι μπορώ να κάνω για να δεχθώ τις ανησυχίες του, αλλά σίγουρα τα δύο σημεία στα οποία αναφέρθηκε είναι σημεία στα οποία είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη και θα δω τι θα κάνω. Για την τελευταία ομιλήτρια για την ενέργεια. Όταν βλέπω τις τροπολογίες δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, είναι αλήθεια. Και σε σχέση με το θέμα της ολοκλήρωσης, πράγματι όταν μιλάμε για μια ολοκλήρωση χωρίς επιπλέον διαιρέσεις θα συμφωνήσω μαζί σας. Για αυτά τα οποία μας είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε, σχετικά με το, το, τις ρυθμίσεις που θα εξυπηρετούν τους πολίτες και όχι τους θεσμούς, Καταλαβαίνω ποια είναι η ανησυχία σας, γνωρίζοντας όμως και αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε εδώ σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα οποία συνειδητοποιούμε και τα οποία είναι δύσκολο να εξηγηθούν στους συμπολίτε μας σήμερα. Όταν βλέπω το πόσο αυξάνεται ε, ο λαϊκισμός διαπιστώνει κανείς ότι το μέγεθος της κρίσης αυτής από την οποία δεν έχουμε εξέλθει καθιστά την εξέταση, την ψύχρεμη της κατάστασης δύσκολη. Και από τότε που ξεκινήσαμε πάλι τις εργασίες μας δεν μπορώ παρά να διαπιστώσω ότι πολλοί από εμά εκφράστηκαν, πήραν το λόγο λέγοντας ότι μπορεί να υπάρξει μια σοβαρή πολιτική κρίση και γι' αυτό ακριβώς καλό είναι να εμείνουμε σε θέσεις και σε ε, απόψεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στις πεπιθήσεις μας προσπαθώντας ταυτόχρονα να είμαστε ευέλικτοι και προσβάσιμοι στους πολίτες μας και να έτσι μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να καταπολεμήσουμε την κρίση όπου λειτουργεί εις βάρος τους. Λοιπόν πρόεδρε, αυτά θα στείλω στους συντονιστές και στους κοιόδης εισηγητές τις συμβιβαστικές μου προτάσεις την Δευτέρα το απόγευμα. Ελπίζω να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε μεγάλη χρονική άνεση και να υπενθυμίσω και την πρόσκληση που απεστάλλει σε όλους έτσι ώστε να δείτε το web doc την Δευτέρα το βράδυ σε μικρές οθόνες τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαδραστικά. Θα παρουσιαστεί το WebDop λοιπόν αυτό την Δευτέρα το απόγευμα στο Στρασβούργο.